So formally, Mrs. European Ombudsman Emily O'Reilly is η Έμιλι Ράιλι, Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, είναι εδώ μαζί μας ε, σήμερα. Θα ακούσουμε με μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον ε, την ε, έκθεσή σας για τις δραστηριότητες του 2014. Συγγνώμη που αργήσαμε, αλλά έπρεπε να συζητήσουμε δύο αναφορές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε για το καλωσόρισμά σας. Δεν χρειάζεται να, καθίστε, να, να, με, να μου ζητήσετε συγγνώμη για την καθυστέρηση γιατί είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Άκουγα την τελευταία μία μισή ώρα online τη συζήτησή σας και με τον κύριο Λεανδίνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν για μένα πάρα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον να ακούω τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε που έχω συζητήσει μερικές φορές μαζί σας και προσφάτως και παλαιότερα. Το γραφείο μου είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να μοιραστούμε μαζί σας τη δική μας εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις μας ε, σε σχέση με όλα αυτά που ε, έχουμε μάθει. Έχουμε και εμείς δυσκολίες, είναι σημαντικό να τις μοιραζόμαστε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα για πρώτη φορά. Το, οι δύο προκάτοχοί μου είχαν ε, πάντοτε εξαιρετική συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών. Είναι η είναι μια από τις πιο σημαντικές επιτροπές και είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Έχουμε την ίδια ε, γραμμή εργασίας. Ε, έχω αυτή την ειδική αποστολή ε, βάσει των συνθήκων και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένας από τους θεσμούς που μας δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, δίνει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχω ρόλο σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Εμένα ε, η δική μου αρμοδιότητα αφορά ε, τα, τις καταγγελίες των ε, πολιτών για τους τα ευρωπαϊκά όργανα και τη λειτουργία τους. Έχουμε πολλά προβλήματα με νομοθετήματα που δεν μεταγράφονται σωστά ή δεν εφαρμόζονται σωστά. Μέχρι τώρα είχαμε μια πάρα πολύ αρμονική συνεργασία και ελπίζω να συνεχίσει. Σήμερα θα σας ε, παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για το 2013. Ε, δεν είναι δική μου δουλειά όμως τόσο, γιατί έχει να κάνει περισσότερο με τη δουλειά του καθηγητή Νικηφόρου Διαμαντούρου, που είναι ο προκάτογός μου και ο οποίος ε, απεχώρησε στις 30 Σεπτεμβρίου. Εγώ ανέλαβα το καθήκον της ε, τελευταίας χρονιάς. Μπορεί να γνωρίζετε κι εσείς ε, ότι κάνω κάποιες έρευνες ε, για να δω που υπάρχουν συστημικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσπαθήσω να κάνω μία αναφορά και σε αυτά. Βασικά όμως σήμερα θα σας μιλήσω για την ετήσια έκθεση για το 2013. Πρόκειται για μία, πρόσφα... για μία μικρή σύνοψη του 2013. Να σας ζητήσω συγγνώμη. Η φωνή μου είναι όχι πολύ καλά. Έχω ένα κρυωματάκι. Ε, πρόκειται για μία σύνοψη η οποία ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα και αφορά με το πώς ε, έρχεται σε επαφή ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με υπαλλήλου που συνταξιοδοτούνται ή που φεύγουν γιατί θέλουν να λάβουν ένα άλλο αξίωμα στον ιδιωτικό, ή να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα. Ο προκάτοχός μου ξεκίνησε τη δουλειά αυτή και εγώ την ολοκλήρωσα. Μία από τις βασικές συστάσεις που έκανα είναι ότι βασίζεται σε δύο ιδέες. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι πράγματι θέλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με ε, πολύ ανοιχτό ε, τρόπο και κατηγορηματικά. Επίσης ελπίζουμε ότι ε, το καθεστώς του προσωπικού δίνει τη δυνατότητα να ε, γίνει κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να ε, επιτύχει αυτό που θέλει, να μην υπάρχουν δηλαδή τόσες φορές περιπτώσεις ε, σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν θα πω πολύ περισσότερα από αυτό, απλώς να πω ότι η βασική μας σύσταση είναι οι ομάδες των ανώτερων υπαλλήλων που θέλουν να φύγουν πρέπει να δημοσιεύονται και πρέπει να γίνεται και μία μικρή αναφορά του ποια ήταν η δουλειά του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια θα είναι η μελλοντική του ε, εργασία στον ιδιωτικό τομέα, να είναι όλα αυτά δημόσια, ώστε να μπορεί να γίνεται μία αξιολόγηση ε, κατά πόσο ε, εφαρμόζονται οι κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων. Υπήρχε μια περίπτωση που ολοκληρώθηκε πέρσι από τον κύριο Διαμαντούρο ε, όταν και αφορούσε το opt-out ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, για την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ήταν ένα τεράστιο γεγονός το οποίο απασχόλησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Νικηφόρος το παρουσίασε και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον κύριο Σούλτς. Αφορούσε την, ε, μια Ιταλική εταιρεία ε, τους ε, είχαν υποσχεθεί ένα ποσό γύρω στα 93.000 ευρώ και τελικά όντως τους δόθηκε το ποσό αυτό. Τον Αύγουστο Άρχισε, ε, ε, δρομολογήσαμε μία ε, εργασία μαζί με τον Νικηφόρο σε σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των agencies. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ συντονίζω ένα δίκτυο ε, συνηγόρων του πολίτη κρατών μελών που ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ανταλλάξαμε πάρα, πολύ, ε, πάρα πολλές πληροφορίες χρήσιμες αλλά και καλές πρακτικές. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω από τότε που ήμουν εγώ ε, συνηγόρος του πολίτη στην Ιρλανδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να ε, μπορούν οι συνήγοροι του πολίτη να είναι σε άμεση επαφή με το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Είναι κάτι το οποίο ανέφερα και τον περασμένο Νοέμβριο ε, το, και αφορά τη Frontex στην Πολωνία και που παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα ασύλου, μετανάστευσης ε, όλων αυτών των ανθρώπων προσπαθούν να ε, έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσουν άσυλο. Η έκθεσή μου ασχολήθηκε με ένα μικρότερης εμβέλειας θέμα ότι η Frontex δεν έχει μια διαδικασία, ε, ένα μηχανισμό καταγγελιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κάτι τέτοιο, ακόμη και αν η ε, καταγγελία πρέπει μετά να ε, διοχετευτεί σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Υπήρχε μια τεράστια υπόθεση που αφορούσε μια παράβαση Είχαν έρθει κάποιοι και μας είχαν πει ότι οι φορολογικές απαλλαγές ε, στην Ισπανία για ορισμένες ποδοσφαιρικές, ε, ποδοσφαιρικούς ομίλους ε, παραβίαζαν το νόμο. Μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να το εξετάσουμε και μας πήρε και πολύ χρόνο να λύσουμε αυτό το θέμα. Λύθηκε τελικά αυτό το θέμα κατόπιν δικής μας παρέμβασης. Άκουσα πάρα πολλά σήμερα το πρωί στη δική σας συζήτηση ότι έχετε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας λόγω των αναφορών που λαμβάνετε, της πληθώρας των αναφορών. Ε, έχουμε ε, με τα χρόνια ε, αναπτύξει έναν πάρα πολύ καλό οδηγό που βρίσκεται διαθέσιμος και στο διαδίκτυο. Είναι ένας χρήσιμος οδηγός για να ξέρουμε πού ακριβώς πρέπει να πηγαίνει κάθε ε, καταγγελία ε, στην Επιτροπή Αναφορών, σε εμά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν πρέπει να λυθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Νομίζω ο κύριος Λιαντίνη τα ανέφερε όλα αυτά σήμερα το πρωί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. 2.400 αναφορές καταφέραμε να λύσουμε ε, πολλές φορές με τη βοήθεια των συνηγόρων του πολίτη. Όταν βλέπει κανείς αυτό το τεράστιο αριθμό, 341 αναφορές ε, αφορούν ε, έρευνες που ξεκίνησαν επί τη βάση καταγγελιών, 461 ε, έχουν ολοκληρωθεί. Φαίνεται μικρός αριθμός αυτός, αλλά ξέρετε οι περισσότερες καταγγελίες ε, καλύπτονται σε επίπεδο κράτους μέλους, και όλες αυτές που αφορούν τα ευρωπαϊκά όργανα θα, είναι, θα έχουν πιο περιορισμένο αριθμό. Όμως το αποτέλεσμα είναι κάποιες ε, έρευνες που γίνονται ούτως ή άλλως. Δηλαδή μία καταγγελία μπορεί να μας δείξει το δρόμο να ε, κλείσουμε και πολλές άλλες αναφορές. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι αυτά τα μικρά νούμερα μπορεί να είναι κάπως παραπλανητικά. Εδώ είναι ο βασικός όγκος των ε, καταγγελιών. Βλέπετε ένα τεράστιο, μια τεράστια στήλη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ότι είναι κακός ε, οργανισμός, απλώς ε, είναι... Οι περισσότερες αναφορές την αφορούν. Βλέπετε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, Γραφείο Επιλογής Προσωπικού, ΕΠΣΟ, ε, είναι ο οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται τις διάφορες ε, αιτήσει πολιτών για εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί. 25,6% ολοκληρώνονται πριν ε, καν γίνουν επίσημες διαδικασίες. Μπορούμε να μιλήσουμε απευθείας ε, με ε, τον οργανισμό και γίνεται μια, ένας φιλικός διακανονισμός κατά κάποιο τρόπο. 43,8% δεν χρειάστηκαν περαιτέρω ε, έρευνες δεν βρέθηκε κακομεταχείριση στις 26, 26% των περιπτώσεων και σε 10,8% των περιπτώσεων βρέθηκε ε, κακοδιαχείριση. Και λοιπές περιπτώσεις 12%. Όσον αφορά τώρα την ε, συμμόρφωση με τις προτάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το, που είχαν γίνει το 2012, κάθε χρόνο γίνεται αυτό και μετά γίνεται μια αξιολόγηση του κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση. Φαίνεται μεγάλος ο αριθμός αυτός, 80% συμμόρφωση και 20% μη συμμόρφωση. Ε, εγώ θα ήθελα να είναι ακόμα υψηλότερο το ποσοστό αυτό σε πολλές ε, ε, χώρες ε, το ποσοστό συμμόρφωση είναι πάνω από 90% το ποσοστό αυτό και αυτή είναι και η δική μου φιλοδοξία, αυτό είναι ο δικός μου στόχος και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν τώρα μεταφέρουμε τις ε, διάφορες ε, υποθέσεις, 52,5% ε, επιστρέφουν στα κράτη-μέλη, κάποια πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13,1% και 37% λυπεί οργανισμοί και φορείς. Εδώ έχετε κάποιες από τις στατιστικές των χωρών. Φαίνεται να είναι πολύ εύβολα τα στοιχεία αυτά, αλλά δεν είναι τόσο. Τεράστιες είναι οι αναφορές που λαμβάνουμε από τους Ισπανούς. Ε, αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κακομεταχειρίζεται τους Ισπανούς, απλώς ε, υπάρχει ένα πάρα πολύ, τοπικό, πολύ, πολύ ε, δραστήριο τοπικό δίκτυο συνήγορου του πολίτη στην Ισπανία και επομένως οι πολίτες γνωρίζουν πολύ περισσότερο ότι μπορούν να έρθουν έρθουν σε επαφή ε, μαζί του ε, για ε, προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. Είναι καλό ότι υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση, ότι γνωρίζουν οι Ισπανοί πολίτες, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα που τελικά την κάνουν διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Γερμανία, Πολωνία και Βέλγιο. Πολλές από τις καταγγελίες ε, προέρχονται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αυτό εξηγεί ε, το γεγονός ότι το Βέλγιο έχει τόσο υψηλό ποσοστό. Δεν είναι οι ίδιοι οι Βέλγοι, αλλά είναι πολλές ε, πολλοί οργανισμοί και πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει που έχουν την έδρα του στι Βρυξέλλε και από αυτού προέρχονται συνήθω οι αναφορέ. Για το Βέλγιο, δούμε μερικά παραδείγματα τώρα το ανέφερα ήδη αυτό, σε πολλέ περιπτώσεις μη κυβερνητικέ οργανώσει ενδιαφέρονται για θέματα δεοντολογίας. Ε, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές καταγγελίες σε σχέση με ισχυρισμούς ε, ε, σύγκρουση συμφερόντων, πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύνθεση ομάδων ενδιαφερομένων stakeholder groups και υπήρχε και μια υπόθεση πολύ επιτυχημένη 140 έγγραφα ε, δημοσιεύθηκαν όταν Γερμανός ε, δημοσιογράφος ζήτησε τα έγγραφα αυτά για την είσοδο της Ελλάδας, ε, στην, την προσχώρηση Ελλάδας στην Ευρωζώνη. μετά βλέπουμε την Ιταλία είναι η εταιρεία που σας ανέφερα προηγουμένως ε, για τα ποσά που τις είχαν υποσχεθεί που τελικά ε, τις δόθηκαν. Στην Ισπανία μίλησα, για την Ισπανία μίλησα προηγουμένως. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίστηκε πολύ κατά πόσο θα έπρεπε να αρχίσει η διαδικασία παραβάση για αυτό το θέμα ή όχι. Τώρα τα βασικά ε, σημεία διαφάνεια, ζητήματα δεοντολογία, συμμετοχή των πολιτών, ε, ε, η πρωτοβουλία των πολιτών που επίσης ήταν αντικείμενο πάρα πολλών αναφορών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά βέβαια στις αναφορές αυτές, προγράμματα που χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κατάλογος συνεχίζεται. Μία ακόμη υπόθεση που ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους. Ε, υπάρχει μία συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που έχουν να κάνουν με σύγκρουση συμφερόντων. Ε, για παράδειγμα, επίτροποι που φεύγουν για να ε, εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις καταλήξαμε ότι δεν υπήρξε πραγματικά σύγκρουση συμφερόντων σε γενικές γραμμές απλώς ε, σε πολλές περιπτώσεις αυτός που πήγαινε ε, να ε, δουλέψει σε στον ιδιωτικό τομέα συνεργαζόταν με μια ένωση δικηγόρων που έκανε ισχυρό λόμπινγκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέτοιου είδους προβλήματα. Πέρσι σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να μεγιστοποιήσω ε, την αξιοποίηση των πόρων του γραφείου μου. 80 άτομα ε, απασχολούνται σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Σκέφτηκα λοιπόν πώς θα μπορούσε το γραφείο μου να είναι πιο χρήσιμο ε, στα ευρωπαϊκά όργανα και συνεπώς και στους πολίτες. Προσπάθησα να εστιαστώ περισσότερο στις τιμικές έρευνες, να εντοπίσω τα θέματα τα οποία ήταν μεγαλύτερου ενδιαφέροντος ε, για τους ευρωπαίους πολίτες. Κάτι το οποίο φάνηκε πολλές φορές που προσπάθησα να χρησιμοποιήσω τους πόρους μου προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε θα ήμασταν πολύ πιο αποτελεσματικοί αν επικεντρωνόμασταν με πιο στρατηγικό τρόπο στο στόχο αυτό. Να χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις, γιατί όπως γνωρίζετε δεν είμαι δικαστής, δεν μπορώ απλώς ε, να επιμείνω να γίνει κάτι. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάνω συστάσεις. Αλλά έχω πάρα πολλές ε, διερευνητικές δυνατότητες και μπορώ να δω οποιοδήποτε έγγραφο, ακόμη και αν είναι πάρα πολύ εμπιστευτικού χαρακτήρα, δεν σημαίνει ότι το δημοσιεύω, αλλά μπορώ να λάβω γνώση του εγγράφου αυτού ή μπορώ να ζητήσω από κάποιον ε, ε, αξιωματούχο να ε, μου παράσχει κάποια στοιχεία. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω όλες αυτές τις δυνατότητες, ώστε όταν κάνω τις συστάσεις μου σε ένα ε, όργανο, να μπορεί να δει ότι είναι πολύ ε, ε, στοιχειοθετημένες και δικαιολογημένες όλες αυτές τις συστάσεις και ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές. τρεις λέξεις που έχουν βαρεθεί να μ' ακούν οι συνάδελφοι να τους λέω. αποτέλεσμα, ε, καταλληλότητα και ορατότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά το θέμα της καταλληλότητας ε, βάσει της συνθήκης του Μάστριχτ ε, έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή αποστολή, είναι σοβαρό καθήκον και οι προηγούμενοι και οι προκάτοχοί μου ε, προσπάθησαν πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και θέλω εγώ να συνεχίσω την προσπάθειά τους. Θέλω ό,τι κάνουμε να είναι χρήσιμο και να έχει αποτέλεσμα να βοηθά ε, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να λειτουργούν καλύτερα αλλά και τους πολίτες ε, να συνεργάζονται και να έρχονται σε επαφή ε, πολύ καλύτερα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό το είπα εν παρόδο, γιατί ο βασικός μου στόχος σήμερα είναι να σας παρουσιάσω την έκθεση για το 2013. Τα περισσότερα σας τα είπα. Η διαφάνεια... Ε, η διαφάνεια και, η, και σε σχέση με την Διατλαντική Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας αλλά και για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ε, προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε και εγώ έχω υποβάλει τις ε, συστάσεις μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορεί να είναι πιο ορατό και πιο διαφανές όλο αυτό. Επίσης ζήτησα από τους πολίτες ποια είναι η δική τους θεώρηση αυτής της διαφάνειας. Θέλω να μου πούν με τα δικά τους λόγια, να μου πούν ακριβώς τι είναι διαφανές και τι δεν είναι διαφανές και για ποιο λόγο θα έπρεπε να είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς δεν ε, κάνουμε. γιατί ακούγονται πάρα πολλές ε, φήμες για το τι έχει συμπεριληφθεί σε αυτήν την ε, συμφωνία, ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες και κάποιοι όχι εγώ δεν έχω ρόλο να διαδραματίσω στην τελική μορφή της συμφωνίας αυτής, αλλά αυτό ο ρόλος που έχω είναι να είναι διαφανής όλη η διαδικασία. Όσον αφορά τη διαδικασία ε, καταγγελιών... Ε, ε, για τα σταλίες έχουμε υπόψη μας την υπόθεση Ασάνς και πολλές άλλες υποθέσεις τέτοιου είδους καταγγελιών είναι πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο θέμα. Οι ευρωπαϊκοί ε, θεσμοί έχουν τέτοιου είδους πολιτική καταγγελιών ε, ε, για να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα για κάποιους όντως να καταγγείλουν μία, να, ε, καταγγείλουν μία ε, ατασταλία, μια, παρατα, μια παρατυπία. Συγγνώμη, να συνεχίσω. Πριν αρχίσω λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία, ε, ήθελα και εμείς να έχουμε στο δικό μου γραφείο τέτοιου είδους ε, πολιτική, γιατί δεν είχε νόημα να το Διατυπανίζω στους υπόλοιπους αν εμείς οι ίδιοι δεν το κάνουμε οι ομάδες επιρρογνωμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πώς ε, ε, συστήνονται, αν υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των επιστημόνων κλπ. Κάναμε μια διαβούλευση, 50 απαντήσεις λάβαμε για το revolving doors, το ανέφερα ήδη αυτό προηγουμένως, και όσον αφορά την πολιτική συνοχής και τα θεμελιώδη δικαιώματα, να υπάρχει ένας μηχανισμός δηλαδή ο, που θα εξασφαλίζει ότι όταν ταπανώνται κονδύλια από τα ταμεία συνοχή στα κράτη-μέλη, τα θεμελιώδη δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν ανησυχίες ότι χρησιμοποιούνται για να ε, γίνονται ε, να γίνονται καταστάσεις περισσότερες για ανθρώπους με ε, αναπηρίες, κάτι το οποίο δεν συνάδει πάντοτε απαραίτητος με το λόγο ύπαρξης αυτών των κονδυλίων. Εγώ προσπάθησα να δω πώς μπορεί ε, να ασχοληθεί καλύτερα η Επιτροπή με το θέμα αυτό και τι ε, σημασία πρέπει να έχει στο ευρύτερο οικοδόμημα ε, των αναφορών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα Φανταστικό το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει και σε σχέση με τους πολίτες για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τεράστιο το έργο αυτό. Πέντε έχουν ζητήσει τον λόγο. Και κυρίως οι αδερφοί. Χάουκε παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Εμιλή που προσήλθατε εδώ η κυρία Άουκεν. Και σε σχέση με την έκθεση Frontex πριν από τις εκλογές το είχαμε εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη, την έκθεση αυτή. Όπως γίνεται όταν εγγράφεται για παράδειγμα μια έκθεση ε, λογοδότησης ε, και αυτό είναι χρήσιμο και παρακολουθώντας τα, πριν φτάσεις εδώ, είχαμε μία συζήτηση για την επίσκεψή μας στη Λαμπεντούζα. Θα το βρίσκες επικοδομητικό αν ε, το εγγράφαμε αυτό και πάλι στην ημερήσια διάταξη διότι σε σχέση με την αντίδρασή μας, σε σχέση με την ε, έκθεση που είχες δώσει στο Frontex, πώς το βλέπεις. Νομίζω μπορούμε να συλλέξουμε διάφορες ερωτήσεις και μετά να τις απευθύνουμε προς απάντηση ε, ώστε να μπορέσουν να απαντηθούν. Προτού φτάσει η ώρα να αποχωρήσετε. Κύριε Μαρία, έχετε τον λόγο. Να σας ευχαριστήσουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην Επιτροπή μας. Ακούσαμε με προσοχή την έκθεση και βεβαίως στη διαδικασία που θα έχουμε εδώ θα τοποθετηθούμε αναλυτικά. Ε, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει βεβαίως και υπάρχει μια σημαντική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, διότι το αντικείμενο είναι να στηρίξουμε ε, να υπάρξει εφαρμογή των δικαιωμάτων και υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Επομένως, είναι ίδια η αποστολή την οποία έχουμε και κατά την έννοια αυτή πρέπει να συνεργαστούμε. Άλλωστε και η στήριξη πολιτική που θα δοθεί από πλευράς Επιτροπής μας στη δραστηριότητα τη δική σας νομίζω ότι είναι κάτι αρκετά θετικό. Θα ήθελα μόνο να σας επισημάνω δύο ζητήματα και θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ε, θα έρθω στο ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες αναφέρετε και είδα και στην έκθεση ότι υπήρξαν και καταγγελίες για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου του Προέδρου της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του κ. Ντράγκη. Η... Το ζήτημα κατά την άποψή μας έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή ο ρόλος της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως μέλη της Τρόικας δημιουργεί αρκετά ζητήματα συμφερόντων. Αυτό το έχει διαπιστώσει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2013. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ε, δραστηριότητά της ως μέλος της Τρόικας ουσιαστικά καθοδηγείται πολιτικά από το Eurogroup, εκπροσωπεί τους δανειστές και έχει αναλάβει να παρακολουθήσει την εφαρμογή των μνημονίων. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλαδή θα πρέπει να αποσκοπεί στην ίδια την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαπιστώσει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μπορεί η Επιτροπή ταυτόχρονα να κάνει δύο δουλειές. Δηλαδή να εκπροσωπεί και τους δανειστές απέναντι σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα να δράει υπέρ του κοινοτικού συμφέροντος. Η σύγκρουση συμφερόντων για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ακόμη πιο σκληρή διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μέλος της Τρόικας υπάρχει εκεί για να, δείχνει, για να δίνει τεχνικές συμβουλές. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι και δανειστής απέναντι σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη, για την Ελλάδα έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομόλογα αξίας 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα αγόρασε αυτά τα ομόλογα με έκπτωση 40%. Κάθε χρονιά όμως απαιτεί να πληρωθούν αυτά τα ομόλογα στο 100%. Και έτσι θα βγάλει κέρδος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εις βάρος του φτωχοποιημένου ελληνικού λαού 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Για φέτος μόνο τα ομόλογα είναι ονομαστικής αξίας 10 δις, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει πληρώσει μόνο 6 δις. Βγάζει λοιπόν κέρδος εις βάρος των πολιτών. Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορούν αυτά τα θεσμικά όργανα να είναι ταυτόχρονα και δανειστές, να είναι εκπρόσωποι των δανειστών και ταυτόχρονα να επιτελούν και τη δραστηριότητά τους ως θεσμικά όργανα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Το δεύτερο θέμα αφορά το κατά πόσο εφαρμόζονται ή πρέπει να υπάρχει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με αφορμή την εφαρμογή των μνημονίων. Διότι προσέξτε υπάρχει μια απάντηση της Κομισιόν προχτές σε συναδέλφους βουλευτές Έλληνες του ΣΥΡΙΖΑ που ρώτησαν αν δεσμεύεται η Κομισιόν κατά τη δραστηριότητά της ως Τρόικα με τα μνημόνια από την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και ξέρετε τι απάντησε. Ότι τα μνημόνια είναι ένας μηχανισμός, είναι κείμενα τα οποία είναι εκτός κοινοτικού δικαίου και δεν υπάρχει υποχρέωση να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα κομμάτι δραστηριότητας και της ίδιας της Κομισιόν που δεν υπόκειται πλέον κατά την απάντηση της Κομισιόν στην τήρηση των θεμελιώδων δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κλείνω με αυτά κύριε Πρόεδρε διότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και εμείς ως Επιτροπή Αναφορών αλλά και εσείς καθώς εξετάζετε τη δραστηριότητα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχετε αυτών των δύο οργάνων. Και θα έλεγα μια πρώτη άποψη αν μπορούσατε να εκφράσετε και ενδεχόμενα αν θα μπορούσατε με βάση αυτά που λέω αλλά μπορώ να σας στείλω και έγγραφα αναλυτικά αν θα μπορούσατε να αναλάβετε μια own initiative report να κάνετε στα θέματα αυτά τα οποία πραγματικά επηρεάζουν την καθημερινή ζωή χιλιάδων πολιτών, πολλών κρατών που είναι σε μνημόνιο όπως των Κυπρίων πολιτών, των Ελλήνων, των Πορτογάλων, των Ιρλανδών κλπ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και το... Now we're proceeding to, to our colleague. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Βαλένσα, συνάδελφο από το ΕΛΚ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αυτή περίπλοκη και σύνθετη θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα. Τον αριθμό των παραπώνων των πολιτών. Κατά το πρώτο έτος έκλεισε περισσότερες εξετάσεις 461 έναντι 350. Μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα θα έλεγα. Επίσης αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν ταχύτατα. 22% έκλεισαν μέσα σε περίοδο τριών μηνών και μετά τα υπόλοιπα μεταξύ τριών και 12 μηνών. Μεγάλο ποσοστό λοιπόν καλύφθηκε μέσα στην περίοδο του ενός έτους. Τεράστιο ποσοστό. Και αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό και θα έπρεπε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα εμείς οι ίδιοι από αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Μια άλλη πτυχή, μια άλλη συνιστόσα. Ποια είναι. Είναι ότι η σωστή διαδικασία όταν υπάρχουν συγκρούσεις και τριβές συμφερόντων και όσον αφορά το θέμα revolving doors, δηλαδή την συνταξιοδότηση ή την στελέχωση με κάποια στελέχη ε, χαίρομαι για το ότι επικεντρωθήκατε με προσοχή σε αυτό το θέμα. Δύο ερωτήσεις θα είχα προς εμάς κυρία ε, Σύνηγορε. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τις μεθόδους που χρησιμοποιήσατε για να μειωθεί η περίοδος ε, όσον αφορά την εξέταση αυτών των χαρτοφυλακίων. Και δεύτερη ερώτηση. Η έκθεση αφορά προτάσεις και μέσα στο πλαίσιο των δράσεων του συνηγόρου κατά το 20% των περιπτώσεων τα θεσμικά όργανα δεν συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις σας. Μπορείτε να μας επεξηγήσετε γιατί, πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο και αν κάτι συμβαίνει ώστε να μπορέσει στο μέλλον να μειωθεί αυτό το ποσοστό. Η κυρία Λεβάση στη συνέχεια. Αλλά μετά θα πρέπει να σας ζητήσω να περιοριστείτε σε ένα 1,5 λεπτό όλοι σας. 1,5 λεπτό. Δεν είναι καλό όταν κάποιος παίρνει το λόγο και δεν σταματάει. Και πρέπει όλοι να αποχωρήσουμε κατά τις 12.30. Έχετε τον λόγο κυρία λοιπόν και μετά θα συνεχίσουμε. Θα είμαστε όμως συντομότεροι στις παρεμβάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, είναι πάρα πολύ αξιόλογη η δουλειά σας. Ε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ανακοίνωσή σας για τα revolving doors, ε, γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε την ακρόαση των υποψηφίων επιτρόπων, ε, μήπως έχουν και εκείνοι σύγκρουση συμφερόντων ε, με το χαρτοφυλάκι που θα αναλάβουν. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν το από πού έρχεται κανείς και πού πηγαίνει. Όλα αυτά τα δύο συνδέονται όταν λέτε ότι πρέπει να ε, για ένα χρονικό διάστημα να ζητούμε από τους ε, επιτρόπους να μην ε, πάνε να δουλέψουν στον τομέα για τον οποίο είχαν αρμοδιότητα, Καλή ιδέα είναι αυτή, αλλά τι θα γίνει όμως, πώς μπορούμε αυτό να το ε, εμποδίσουμε και να το περιορίσουμε όταν ε, οι υπάλληλοι που δούλευαν ας πούμε σε ένα βιομηχανικό τομέα, πώς θα, σε ένα συγκεκριμένο τομέα, πώς είναι δυνατόν να τους εμποδίσουμε από το να πάνε μετά να δουλέψουν σε έναν τομέα για τον οποίο είχαν αρμοδιότητα. Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να το κάνουμε αυτό. Όσον αφορά τώρα ε, τη δήλωση συμφερόντων. Την ΕΦΣΑ, α πούμε, εμείς ε, την κατακρίναμε ή κάποια μέλη της Επιτροπής Μπαρόζο. Ε, πρέπει να είμαστε πραγματικά δρακόντιοι ε, ως προς τη δήλωση συμφερόντων για ανθρώπους που δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή είναι για παράδειγμα επιστημονικοί σύμβουλοι. Υπάρχει το εμπορικό απόρριτο για να το πω έτσι. Εγώ επειδή είμαι εισηγήτρια για ένα τέτοιο θέμα και μιλάω για το θέμα της διαφάνειας στον βιομηχανικό τομέα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα επιμείνω πολύ. Η Όλαφ επίσης που είναι ο οργανισμός καταπολέμησης απάτης. Πάρα πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας ζητήσω εσάς συγκεκριμένα να, ε, να ζητήσετε από την Όλαφ να μας πει ακριβώς τι κάνει γιατί ναι, με λαμβάνουμε μια έκθεση, αλλά μετά δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφάνεια σε συνέχεια μια καταγγελία που εμεί κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο τη διαφάνεια των ε, υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η Σα ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντα για το έργο το οποίο επιτελέστηκε από την συνήγορο μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έργο που έδειξε μεγάλη δραστηριότητα και αποτελεσματικότητα. Κυρίως θέλω να συγχαρώ και την συνήγορο για την έρευνα που έκανε και ιδιαίτερα για το, τη θεματολογία που ήταν πολύ κοντά στη θεματολογία που οι πολίτες απασχολούνται με αυτήν και σε σχέση με τις ε, κλινικές ε, δοκιμές για παράδειγμα έκανε τα πειράματα δηλαδή έκανε έργο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα ενδιαφέροντα των πολιτών και τα αιτήματά τους. Μεγαλύτερη, ε, πιο ευδιάκριτος χαρακτήρας υπέρ του έργου που επιτελείται από το συνήγορο ή τη συνήγορο του πολίτη και πραγματικά να δούμε πώς είχε αυτή η διαδικασία ώστε να μπορέσει να δρομολογηθεί η βελτίωση του ευδιάκριτου του χαρακτήρα αυτού του έργου που μας ενδιαφέρει και εμάς στην Επιτροπή Αναφορών για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια μεγαλύτερη διείσδυση και του δικού μας έργου. Και μια απλή ερώτηση που αφορά το θέμα του αν θα το εξετάζατε εσείς ε, ως ε, ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Τι γίνεται σε σχέση με αυτή τη σημαντική κρίση που είδαμε και είδαμε πώς τα διάφορα κράτη-μέλη ε, προσπάθησαν ή ε, αντιμετώπισαν τον πειρασμό να ερμηνεύσουν διαφορετικά διάφορα πράγματα σε σχέση με το πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, τα θέματα όπως για παράδειγμα την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και ιδιαίτερα την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Θα το θεωρούσατε σημαντικό να αναλυθεί το πώς η κρίση και η αντιμετώπιση της κρίσης είχε επιπτώσεις στην ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων και πώς αυτό ε, υπέστη ε, κάποιες επιπτώσεις ε, σε σχέση με το κυρίαρχο αυτό δικαίωμα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κυκλοφορούν ελεύθερα. One, Ευχαριστώ. Έχω τώρα τέσσερις ακόμα ευρωβουλευτές ε, στον κατάλογο. Μπορούμε να κλείσουμε μετά από αυτά τα ονόματα της παρεμβάσεις στον κατάλογο. Εξαιρετικά. Η κυρία Βαλίνα παρακαλώ. Sí, Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη συνήγορο των πολιτών, κυρίως για αυτή την ειδική έκθεση και αυτή την πρωτοβουλία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, που ήταν η ειδική έκθεση για τις απάτες. Σε αυτή την ε, έκθεση αυτού του τομέα υπάρχουν στοιχεία τα οποία παραβιάζουν τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ξέρω ότι η προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ήταν κάτι στην οποία δεν συντάχθηκε η έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως επειδή βρισκόταν στο τέλος της ε, εντολής της ε, και δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Θα ζητούσα λοιπόν μια και έχει τέτοια σπουδαιότητα και παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα μυριάδων πολιτών σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία πραγματικά να συνταχθεί αυτή η έκθεση από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you. Now the floor is to Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζάκη νομίζω, ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ. Τσάκι είναι η σωστή προφορά, αλλά δέχομαι και άλλου είδους ε, εκφορά του ονοματός μου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία για την παρουσίασή σας και ιδιαίτερα για το έργο σας ε, όπως αναφέρθηκε και σε σχέση με, και με τη Σλοβακία βλέπω αυτό το χάρτη τώρα που είναι πολύ χρήσιμος για όλους μας ε, και κάπως εκπλήσωμαι για τη χώρα μου εδώ βλέπω ότι κάποιες αποδεκτές περιπτώσεις έχουν ε, αντιμετωπιστεί, αλλά είναι μηδέν, μηδέν ο αριθμός για τις, ε, ε, ε, τα αιτήματα αυτών των πολιτών. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Ελπίζω ότι δεν είναι μια αρνητική διακριτική αντιμετώπιση ή μεταχείριση των πολιτών μιας μικρότερης χώρας. Και γραπτός θα μπορούσατε ίσως να απαντήσετε ή με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα μπορούσατε να μου αποστείλετε αν χρειαστεί. Η κυρία Μπεατρίς Μπεσέρα παρακαλώ έχει τον λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Ρέλη για μια εξαιρετική έκθεση, για έργο, δουλειά ιδιαίτερα σπουδαία σε αυτό το ε, χρόνο που εργάζεστε κυρίως για ένα θέμα στο οποίο νομίζω μεταφράζονται όλα τα ε, θέματα αυτά. Ο υποδειγματικός ρόλος, υποδειγματικός χαρακτήρας ότι από πλευρά συνήγορου του πολίτη υιοθετείται μια τέτοια προσέγγιση είναι το πρότυπο που πρέπει να ακολουθηθεί. Και είναι το πρότυπο για αυτά τα στοιχεία που έχουν σημασία μεγάλη όπως είναι η διαφάνεια όπως είναι η διασφάλιση ανεξαρτησίας και μη σύγκρουσης συμφερόντων. Και ο υποδειγματικός χαρακτήρας είναι εκείνο το οποίο δίνει νόημα στο έργο μας και θα επιτρέψει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια και να διασφαλίσουν στους πολίτες που εμείς εκπροσωπούμε ότι όταν συμβαίνει κάτι έξω από τα όρια στα οποία θα έπρεπε να συμβαίνει, θα πρέπει αμέσως να δραστηριοποιούμαστε για να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι η βαθύτερη έννοια σε σχέση με το έργο σας. Απλά μια ερώτηση θα ήθελα να σας υποβάλω και να την τοποθετήσω σε σχέση με τις προτεραιότητες ε, στις οποίες αναφερθήκατε και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτές. Μια παρατήρηση απλά θέλω να κάνω σε σχέση με κάτι που υπογραμμίσατε και τονίσατε ο μεγάλος αριθμός 1 ως περίπτωση της Ισπανίας για τον μεγάλο αριθμό αναφορώ και παραφώνων, παραπώνων που συντάσσονται και αποστέλλονται από Ισπανούς υπηκόους σε σχέση με την Ισπανία. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτός ο ευδιάκριτος χαρακτήρας και αυτή η σπουδαιότητα όλων αυτών θεωρείται ότι υπάρχει κάποια βελτίωση που πρέπει και μπορεί να γίνει και να επιτελεστεί θα ήταν κάτι το οποίο θα διευκόλυνε το ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους ε, και σε σχέση και με το όργανό σας το οποίο ασχολείται με αυτά τα θέματα, να επικεντρώνεστε σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα παρακαλώ έχει τον λόγο τώρα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κυρία Ορέλη για το έργο σας κατά το παρελθόν ε, έτος που διέτρεξε για να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ένα σχόλιο που θα ήθελα να αναφέρω και αυτό αφορά τη σελίδα 29, το 20% της ε, απουσίας συμβατότητας ή ε, ευθυγράμμισης. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω για τις απόψεις ώστε να μειωθεί κατά το άμεσο μέλλον αυτός ο αριθμός, αυτό το ποσοστό. Σας ευχαριστώ. Αυτό ολοκληρώνει τον κατάλογό μου. Έχετε τώρα τον λόγο κύριε Ορέλη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις έγιναν και σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις καλύψω, να τις απαντήσω και να με συγχωρήσετε αν υπάρξουν κάποια κενά. Αλλά το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό για εσάς ώστε να δοθεί συνέχεια σε αυτά. Κυρία Όγκεν, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για το γραφείο μας να υπάρξει αυτή η τοποθέτηση και δραστηριοποίηση. Σπάνια υποβάλλεται μια τέτοια έκθεση όσον αφορά το Κοινοβούλιο για να υπάρξει ειδική δραστηριοποίηση. Και καλό είναι να μπορεί να προσέρχεται ε, όταν προσέρχεται υπερβολικά συχνά κάποιος στο κοινοβούλιο ίσως δείχνει ότι κάτι δεν ε, πάει καλά. Όταν έρχομαι εγώ στο κοινοβούλιο πραγματικά θέλω να δείξω ότι χρειάζεται αυτή η υποστήριξη. Για την έκθεση αυτή κάπως με τις εκλογές ίσως ε, ας το πω έτσι απολέστηκαν ε, αρκετά στοιχεία και είχε, υπήρχε ειδικό βάρος νομοθετικού έργου, για το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να μπορέσει να περάσει και να συζητηθεί στην Ολομέλεια αυτό το ε, στοιχείο, αυτή η έκθεση γιατί έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Είναι μικρό, ας το πω έτσι, μικρής, μικρό έγγραφο στην έκθεσή του αλλά έχει μεγάλη σπουδαιότητα και μας αφορά όλους και τους πολίτες υπό την πτυχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κυρίε Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ και για τα ευγενικά σας λόγια για τη συνεργασία όπως θα έπρεπε να διασφαλιστεί. Και ουσιαστικά ε, αναφέρεστε και στοχεύετε στο ίδιο και είναι σημαντικό αυτό. Σε σχέση με την παρέμβασή σας, αυτό που ανείχνευσα είναι ότι υπάρχει κάποια απογοήτευση από εσά και αντανακλά και κάποια απογοήτευση πολλών πολιτών και άλλων στην Ελλάδα σε σχέση με την Τρόικα και που κάποιοι είδαν ως απουσία λογοδότησης ή ε, απόδοσης ευθυνών διότι δημιουργήθηκε ένα ε, αξιοπερίεργο όν που ε, συναποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Ποιο ήταν τελικά δηλαδή αυτό το ε, μόρφωμα. Προέρχομαι από μια χώρα που αντιμετώπισε την Τρόικα επί μια σειρά ετών και γνωρίζω αυτό το ζήτημα συγκεκριμένα. Ως συνήγορος, όταν κάποιος προσέχεται σε μένα με οποιοδήποτε ζήτημα, θα ε, ε, προσπαθώ να δω πού θα μπορούσε να υπάρξει ρεαλιστικά η δική μου πιο αποτελεσματική εμπλοκή για να υπάρξει και το μέγιστο αποτέλεσμα. Αλλά συνειδητοποιώ απόλυτα και το πολιτικό, πολιτικού χαρακτήρα ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε. Συνέταξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ειδική έκθεση για τη δράση της, ε, δράση της Τρόικας στην Ελλάδα. Και βλέποντας, ανασκοπώντας ε, τη σύνθεση και το πώς λειτουργήσε η Τρόικα, πολλοί αναγνώρισαν ότι υπήρξαν κενά και ανεπάρκειες ε, στη δράση της. Και είδαν οι πολίτες ε, δημοκρατικό έλλειμμα, απουσία δημοκρατικής δράσης στο πώς λειτουργήσε η Τρόικα. Και αυτό οδήγησε σε πάρα πολύ πιεστικές καταστάσεις ε, σε κρίσιμες περιόδους. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσα να έχω τα στοιχεία αυτά και σε ένα διάλογο μαζί σας να δω πώς μπορώ να εμπλακώ με εποφελή τρόπο και να χρησιμοποιήσω τις εξουσίες και αρμοδιότητες μου πιο εποφελώς. Ε, ιδιαίτερα εκτιμώ θετικά το πλαίσιο αυτό μεταξύ ε, πολιτικών ε, και των ε, δραστηριοτήτων του δικού μου γραφείου. Κύριε Βελάθκε, θα ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε να έχουν τις ύψιστες, υψηλότερες προδιαγραφές λειτουργίας τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και υψηλές προδιαγραφές κάποια κράτη-μέλη σε συγκεκριμένα θέματα. Στην αποτελεσματικότητα ως ζήτημα είναι ένα πλήρες, ένα ε, περίπλοκο θέμα για, το, για τα κενά που υπάρχουν, ε, βάρος, ε, άρθος παρελθόντος κτλ. Και σε σχέση με τα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο συζητάμε. Ένα ιδιαίτερο εγχείρημα στο, με, το δικό μου αξίωμα στην Ιρλανδία προσπάθησα να ακολουθήσω όταν είχαμε τη μελέτη Time and Motion, βλέποντας δηλαδή τις δομές ε, και μετά αποσυναρμολογώντας τα στοιχεία να τα ανασυνθέσουμε με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κάτι το οποίο είναι κοινό σε εκείνους που προσπάθησαν και πέτυχαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους είναι αυτό. Και αυτό κάνουν από τη στιγμή που φτάνει ένα παράπονο ή μια αναφορά. Είναι θεμελιώδους ε, χαρακτήρα, είναι τεράστια σπουδαιότητα να γίνεται αυτό έγκαιρα και άμεσα. Τα παράπονα, οι προσφυγές, οι αναφορές που ε, φτάνουν στα χέρια μας να είναι αποδεκτές και αποδεκτά. Και αν ε, ενταχθούν πόροι σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το σε αυτή την πρώτη φάση στην αλυσίδα των δράσεων αυτό μπορεί να πετύχει πολλά στο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα Στη συνέχεια σε επόμενη παρέμβαση για την ανακύκλωση στελεχών, revolving doors και κάποιους υπαλλήλους, πρώην υπαλλήλους που αναλαμβάνουν ε, δραστηριότητες που συγκρούονται με τα προηγούμενα καθήκοντά τους, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, κατά τη διάρκεια της δράσης μας για την εξέταση της κατάστασης των ανακυκλώσεων Πρώτον, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά υπαλλήλους, για παράδειγμα, ε, που μπορούν να υπάρξουν περικοπές όσον αφορά και τις συντάξεις τους, όσον αφορά κάποιους, ε, κάποιες περιπτώσεις. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με πρώην επιτρόπους, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και με αυτούς. Ε, αυτό στο οποίο προσπάθησα να επικεντρώσω το δικό μου έργο τις δικές μου κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς και συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού του θέματος είναι να πούμε ότι ο ήλιος, οι ακτίνες του ήλιου, το φως του ήλιου είναι το καλύτερο απολυμαντικό. Και έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει διαφάνεια διότι αυτό είναι αποτελεσματικό, διότι δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να απολυθεί ε, ο οποιοδήποτε. Αν όμως οι κυριότεροι, οι υψηλοί αξιωματούχοι θα γνωρίζουν ότι όταν θα περνάνε στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να υπάρχει μία περίοδος χρονική, όχι μόνο να πούν στην Επιτροπή που θα πάνε, αλλά και να μην αναλάβουν τέτοια καθήκοντα για συγκεκριμένο διάστημα, αν αυτό είναι ευδιάκριτο για τους πολίτες και υπάρχει γνώση ότι η Επιτροπή θα εξετάσει ακριβώς ε, και θα επιβάλλει εκείνες τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν, ε, τότε αυτό θα επιτρέψει σε άτομα όπως η Μάσα ε, ή και για άλλους ε, να βλέπουν και να εποπτεύουν το τι συμβαίνει και αυτό θα έχει επίπτωση στο πώς θα φέρεται ο καθένας και τι θα κάνει. Πιστεύουμε ότι τα νομικά μέσα και δυνατότητες μέσω του κανονισμού των υπαλλήλων υπηρεσιακού κανονισμού υφίστανται αυτά τα μέσα ήδη και υπάρχουν. Αλλά πέρα από αυτό και σε αυτή τη διαδικασία επιβολής ε, ε ποινών ή προστήμων ή κυρώσεων και αυτό θα ενδυνάμωνε αυτή την προσπάθεια. Και αν υπάρχουν κάποια παράπονα φυσικά, ε, τότε φυσικά ε, θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Τώρα, σε σχέση με την επόμενη παρέμβαση που έγινε, τη Δευτέρα θα έχουμε την ε, ε, διασφάλιση του διεθνούς δικαιώματος να μπορεί κανείς να έχει γνώση συγκεκριμένων πραγμάτων και σε σχέση με τα ε, κλινικά στοιχεία και επιστημονικά στοιχεία για πειράματα και τα λοιπά θα υπάρξει παρέμβαση και από την Ευρωπαϊκή Αρχή των, για την Ιατρική και επαΐοντες που είναι πολύ καλά γνωστοί και ε, γνωρίζουν το θέμα θα μπορέσουν να παρέμβουν. Από πλευράς άλλου Ευρωβουλευτή αναφέρθηκε το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της Frontex. Ένα από τα θέματα που με απασχολούν είναι ως συνήγορος του πολίτη να προσπαθώ να μεγιστοποιήσω το δυναμικό και την αποτελεσματικότητα ε, στην Ευρώπη. Εξετάζω να βρω πού θα υπάρχουν το μισο που θα μπορούσα να κάνω κοινέ εξεταστικές έρευνες ή διακριβώσεις με τα κράτη-μέλη και τους ε, αξιωματούχους τους ώστε να γίνει κάτι πιο αποτελεσματικό. Εξετάζω ιδιαίτερα λοιπόν τις δυνατότητες που ε, μπορούν να αναφύονται στον τομέα τομέα της Frontex και σε σχέση με τη μετανάστευση και τους μετανάστευς. Μετανάστες. Για σας κύριε Τσάκη, για τη Σλοβακία που αναφέρατε, 31 περιπτώσεις στο μηδέν, από 31 περιπτώσεις σε μηδενικό ε, επίπεδο. Αυτό όχι επειδή αγνοούμε με κανένα τρόπο την ε, Σλοβακία, αλλά βρισκόντουσαν εκτός πλαισίων που θα μπορούσαμε εμείς να δραστηριοποιηθούμε για να εξετάσουμε. Έτσι λοιπόν ε, μπορείτε τουλάχιστον να δείτε τι έγινε σε κάθε ε, περίπτωση στο έργο μας. Από πλευράς άλλου Ευρωβουλευτή έγινε παρέμβαση για ε, θέματα διαφάνειας και σύγκρουση συμφερόντων. Και την Ισπανία είναι ένα θέμα που όταν έχουμε ε, διάφορους συνήγορους πολιτών ε, που συνέρχονται υπάρχει πάντα συζήτηση γιατί στη Δανία να πούμε ή σε κάποιες άλλες χώρες ή στην Ιρλανδία για παράδειγμα για το δημόσιο τομέα για παράδειγμα έχουμε αναπτύξει μια, ε, μια σειρά τομεακών συνηγόρων για τη βιομηχανία της επιχειρήσεις, για τα παιδιά, για τις συντάξεις και για έναν άλλο τομέα που ε, διέλαθε τις προσοχής, ε, ε, διαφεύγει της προσοχής μου αυτή τη στιγμή. Κάθε χώρα λοιπόν, κάθε κράτος μπορεί να αποφασίζει αυτοδίκαια και αυτοτελώς ποιες ανάγκες υπάρχουν και τι θα προτιμούσε να κάνει και πώς. Τα πιο σημαντικά όμως από πλευράς κάθε χώρας είναι να επιλέγονται οι δυνατότητες που δίνουν αποτελέσματα και σε σχέση με την, τον πολλαπλασιασμό συνηγόρων αυτό δημιουργεί και σύγχυση στο τέλος τέλος για τους πολίτες. Δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορές ποιότητας στα επιτεύγματα ή στα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη δράση ε, διαφορετικών συνηγόρων. Το πιο αποτελεσματικό είναι να δούμε τι είναι το πιο αποτελεσματικό, πιο εξορθολογισμένο και πιο ε, ορθολογικό ε, ώστε να μπορέσει να ε, προτιμηθεί και να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά. Ματσόλα, ναι. Κάνατε λόγο για το 20% έτσι δεν είναι, για τις συστάσεις ε, από πλευράς μας. Και σε σχέση με τα όσα δεν έτυχαν συνέχεια, το 80% και αυτό μας ανησυχεί αυξάνει για το 20% μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Δεν μπορεί να μην υπήρξε κάποια συμφωνία και διάφοροι άλλοι λόγοι. Εκείνο όμως που ελπίζω ότι θα μπορέσω να πράξω είναι να μπορέσω να ε, βελτιώσω το πώς συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποστέλλονται επιστολές. Εμείς αποστέλουμε μια επιστολή προς αυτήν, εκείνοι απαντούν με επιστολή. Εγώ θα ήθελα μια πολύ πιο άτυπη σε κάθε επίπεδο επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα μέσω προσωπικών επαφών που θα βελτιώσουν τα πράγματα. Και κατά την ε, έναρξη της ανάληψης των καθηκόντων μου ή σύντομα μετά έδωσα ιδιαίτερη σημασία να συνέθω με το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσουμε μια μικρή ομάδα με δικούς μου αξιωματούχους και αξιωματούχους τους ώστε να δούμε για τα πιο σημαντικά προβλήματα ποια λύση θα μπορούσε να επιλεγεί και να στοχεύσουμε σε αυτή. Ήθελα να, να δείξω το πνεύμα συνεργασίας και προθυμίας δεν μπορώ να επιβάλλω σε κανένα απόψεις ή δράσεις, αλλά είμαστε ένα πραγματικά ανεξάρτητο, ε, ανιδιοτελές και θα έλεγα χωρίς να ε, υπάρχει οποιαδήποτε ανάμειξη όργανο και σε σχέση με τις συστάσεις ε, και τις δράσεις μας θα πρέπει να εξευρεθεί και ο σωστότερος τρόπος για να υιοθετηθούν τα αναγκαία μέτρα από άλλα θεσμικά όργανα αν δράσουμε προς όφελος αυτής της κατεύθυνσης όλοι μας, τότε αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήσασταν ε, σήμερα εδώ και απαντήσατε ε, σε όλους μας τους συναδέλφους, ονομαστικά μάλιστα, τις ερωτήσεις που σας έθεσαν. Είναι δύσκολο να συλλάβουμε το μήνυμα, αλλά η ο αντίκτυπος, ε, η απόδοση και η διαφάνεια είναι οι τρεις βασικές λέξεις ε, και όλοι μας προσβλέπουμε σε βελτιωμένη και περισσότερη συνεργασία μαζί σας σε διάφορους τομείς. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ όλους συνάδελφοι. Τα ξαναλέμε στις 3 το απόγευμα.